θεωρώ ότι είναι ευπρόσδεκτη αυτή η προστασία, η οποία εναρμονίζει τις διατάξεις για την προστασία των καταγγελώνων σε όλα κράτη-μέλη, γιατί σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπήρχε τέτοιου είδους προστασία. Θέλουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο να προστατεύεται. Η παραβίαση του νόμου είναι Πραγματικοί υπάρχουν φορολογικές παραβιάσεις, ε, παραβιάσεις σε βάρος των Ευρωπαϊκών Ταμείων και αυτοί που αναφέρουν τα θέματα αυτά κάνουν πολύ σημαντικό έργο. Υπάρχουν όμως μέσα που θα πρέπει να επιτρέπουν η προστασία να είναι ουσιαστική. Καταρχήν χρειαζόμαστε εμπιστευτικότητα, αλλά θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε την ε, προστασία και στην άλλη, της άλλης πλευράς των κατηγορουμένων ε, για παρατυπίες, διότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και την κακόβουλη καταγγελία. Και αυτή η γραμμή είναι πολύ λεπτή, δεν θέλουμε να παραβιάζεται. Με τα χαράς λοιπόν θα ήθελα να προτείνω να σκεφτούμε και την άλλη πλευρά όταν θα υλοποιηθεί αυτό. Ευχαριστώ. Ε, έκθεση κλίντς, διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων. Συνεχίστε κύριε Πόλτσακ. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων είναι σαφής, σαφώς σημαντική για την Ευρώπη. Η νομοθεσία αυτή μπορεί να μην είναι ιδανική, σε βάση των όσων λένε οι συνθήκες ότι μπορεί να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σαφώς είναι μια πρώτη διαμεθοριακή προσπάθεια για την προστασία για τα κεφάλαια αυτά. Πρέπει να υπάρχουν ίσες ε, συνθήκες για τις επιχειρήσεις, αφαίρεση των εμποδίων για την ελεύθερη διακίνηση, ας πούμε, μετοχών, με στόχο τη δημιουργία ενός ε, δίκαιου ε, πεδίου αλλά πρέπει να υπάρχει καλή προστασία και να επιτρέπεται στους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν το ελεύθερο κεφάλαιο τους. Χαίρομαι που οικοδομούμε μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, την οποία πολύ υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι. Η έκθεση Wolf Klintz, διασυνορική διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων. Ευχαριστώ. Όλο και περισσότεροι ε, εξοικονομούν χρήματα, αποταμιεύουν χρήματα για επενδύσεις και επενδυτικά ταμεία και επενδύουν σε μετοχές που θεωρούν ότι έχουν δυνατότητες. Αυτό είναι ουσιαστικά καλό. Είναι καλό που όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναλαμβάνουν προσωπικά την ευθύνη τους και δεν υπάρχουν ε, ε, μόνο επενδυτικές επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους. Αλλά υπάρχουν και διάφορες προκλήσεις από αυτή την ελεύθερη ε, διακίνηση του κεφαλαίου, κυρίως για το κεφάλαιο αυτών των ανθρώπων που αποτολμούν να μπουν στη ζούγκλα της ατομικής επένδυσης. Χρειάζεται λοιπόν κάποια προστασία για την παροχή εγγυήσεων στους ιδιώτες επενδυτές η οδηγία αυτή εν μέρη το εξασφαλίζει και όχι δεν το εξασφαλίζει επαρκώ και γι' αυτό δεν την υποστήριξα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλη έκθεση, Σέμον. Κύριε Μέσσερ Σμιτ, έχετε το λόγο. Κεφαλαϊκέ απαιτήσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο γιατί ήθελα να αναφερθώ στο γενικότερο πρόβλημα που έχουμε, το γενικότερο θέμα που έχουμε σε αυτόν τον τομέα συμφωνήσαμε ε, να φτιάξουμε κάποιους κανόνες μαζί για την ελεύθερη οικονομία, για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων κτλ. Ε, ειδικότερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά υπάκουοι στα όσα λένε οι διάφορες αρχές ε, οι Αμερικανοί. Δεν δέχονται οδηγίες που δεν ε, προσαρμόζονται στο αμερικανικό μοντέλο. Εμείς ε, στη Δανία αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε πράγματα που αφορούν τη δική μας περίπτωση. Πρέπει λοιπόν να ε, διασφαλίσουμε ότι το επόμενο κοινοβούλιο θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά με τα όσα γίνονται στην Επιτροπή αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην περίπτωση αυτή υπερψήφισα και θα εξηγήσω γιατί. Εξακολουθούμε να νιώθουμε τα, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 2007-2008. Δεν έχουν ακόμα επιληθεί όλα τα προβλήματα της σταθερότητας των ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτων και δεν έχουμε μειώσει τους κινδύνους στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχουμε όμως μελετήσει την καθαρή χρηματοδότηση του συστήματος. Συμφωνώ με τα μέτρα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο ώστε να είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες καθώς και η μετάδοση των πληροφοριών για όσους συμμετέχουν στον χρηματοοικονομικό τομέα. Θα ήθελα να εξηγήσω τι θα επιφέρει αυτό. Πρόκειται για κάτι το πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σκέλη. Εγώ ψήφισα υπέρ των κεφαλαϊκών απαιτήσεων και τη σχετική οδηγία ε, ώστε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα μέτρα που προτείνονται για το μετριασμό των κινδύνων θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις για τα αγαθά και τις υπηρεσίες και θα ενισχύσουν την αντοχή των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι απαιτήσει για τι μικρότερε τράπεζε ε, θα επηρεάσει ε, θετικά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Υποστηρίζω πιο ευέλικτε ε, προποθέσει για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, Υποστηρίζω την ανάπτυξή του. Πρέπει να μεταχειριζόμαστε τι μικρομεσαίε τράπεζε, τι μικρέ τράπεζε αναλογικά. Υποστηρίζω την εστίαση στην ευαισθησία στους κινδύνους ώστε να δημιουργήσουμε ε, σταθερότητα και μια στιβαρή ευρωπαϊκή οικονομία μετά την κρίση. Εδώ έχει επιτευχθεί μια καλή ισορροπία μεταξύ τη μείωση των κινδύνων και τη συνέχιση τη ενθάρρυνση ε, τη χρηματοδότηση και των επενδύσεων. Ο κύριος Σιμών και οι συναδελφοί του έκαναν πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη έκθεση, Φερνάντεθ. Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο, παρακαλώ. Τα ομόλογα που είναι διασφαλισμένα με κρατική εγγύηση είναι ένας μηχανισμός ο οποίος βεβαίως δεν μπορεί να αριθμίσει τις, τα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία της ε, ευρωζώνης. Θα πρέπει καταρχάς να υπάρξει θεσμοθέτηση των ευρωομολόγων από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ποσοτικής χαλάρωσης. ο κύριος ντράγκη παρανόμως έχει αποκλείσει τα ομόλογα τα κρατικά τα ελληνικά από την ρύθμιση της ποσοτικής χαλάρωσης. με τον ίδιο τρόπο έχει επίσης αποκλείσει και τα ομόλογα των εταιριών των ελληνικών εταιριών από την ποσοτική χαλάρωση. αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυξημένη ρευστότητα στην ίδια την ελληνική οικονομία μια οικονομία που διαλύθηκε από την τρόικα. ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες ρυθμίσεις προκειμένου χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα όπως η ελλάδα να μπορούν να ανασάνουν. γι' αυτό το κίνημά μας ελλάδα ο άλλος δρόμος προτείνει να υπάρξει μια ειδική σχέση της ελλάδας με στην ευρωπαϊκή ένωση και στην ευρωζώνη. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Άλλη έκθεση. Κάρας Μπερές για τα χρηματοδοτικά μέσα. Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης. Κύριε Κέλλη, έχετε το λόγο. Sorry. Υποστηρίζω τις τροπολογίες αυτές ε, για την οδηγία αυτή, την εισαγωγή πιο προχωρημένων εργαλείων, ε, οι πλατφόρμες κοινοποίηση ε, και ενημέρωσης, ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές και τις εποπτικές αρχές και τις εθνικές αρχές. Μερικά από τα προτινόμενα εργαλεία είναι αυτά για τη σύγκληση και τη συνεργασία στον τομέα των ασφαλίσεων. Είμαι υπέρ αυτής της προσέγγισης που εστιάζεται στους καταναλωτές όσον αφορά την εποπτεία, βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ κρατών μελών και αναφορά στοιχείων από τους παρόχους για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Υποστηρίζω την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις ασφαλίσεις στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεχόμενη ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε θέματα χρηματοοικονομική εποπτείας, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ισορροπία στι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Αρχής ε, ασφαλισίων και επαγγελματικών συντάξεων και των εθνικών αρχών. Ε, πολύ καλή ισορροπία εδώ επιτεύχθη. Ε, συγχαρητήρια στον κύριο Καρέσκη και την κυρία Μπερέ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Θα έχετε ξανά το λόγο τώρα για την επόμενη έκθεση. Φέρμπερ, προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων και επενδύσεων. Παρακαλώ, κύριε Κέλλη. Okay, To... Συγχαρητήρια πάλι στον συνάδελφο Μαρκούς Φέμπερ. Οι κανόνες που αφορούν τις επενδυτικές εταιρείε ε, ε, είναι καλοί και πρέπει να αντιμετωπιστούν οι σχετικοί κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα όταν η κλίμακά τους είναι τέτοια που οποιαδήποτε αποτυχία τους δημιουργεί συστημικό κίνδυνο για την οικονομία, διότι οι επενδυτικές εταιρείε ε, έχουν μεγαλύτερα, πιο επικίνδυνα ανοίγματα από τις τράπεζες και πρέπει να δρουν πιο οργανωμένα. Οπότε έχει νόημα να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι και δεν μπορούν να ε, εφαρμοστούν ε, σε αυτές οι ίδιοι κανόνες. Η εφαρμογή διαφορετικών κανόνων για μικρές μη συστημικές εταιρείες θα βοηθήσει επίσης να βελτιωθεί η διαφάνεια και να παρασχεθούν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εμπιστοσύνη στις επενδύσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνεται από τα επενδυτικά ταμεία με την εισαγωγή κανόνων προσαρμοσμένων στο επιχειρηματικό μοντέλο τέτοιων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση. Η κυρία Σόιτροβα. Διαφανής και προβλέψιμη ώρα εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που η οδηγία εγκρίθηκε και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία η διαφθηνής και προβλέψιμη ώρα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική και για εργοδο... τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους, ώστε να τους παρέχει βεβαιότητα για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν σε πιο χρονικό διάστημα όταν ε, είσαι εργοδότης και για τους νέους εργοζόμενους και για τους υφιστάμενους. Η συμφωνία στο πελαίσιο του τριμερούς διαλόγου είναι αρκετά ισορροπημένη και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους και γι' αυτό υπερψήφισα. θα, θα ενημερώνονται νωρίτερα οι εργοδότες για τα δικαιώματα ως οι για, τα, ε, δικαιώματά τους. Η τελική διατύπωση σέβεται την εθνική νομοθεσία που μπορεί να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις τοπικές ιδιαιτερότητες της αγοράς χωρίς να αποτελεί μεγάλο διοικητικό άχθος για τους, αγορ... Ε, για τους εργοδότες που είναι σοβαρό. Ευχαριστώ κύριε Στροεύσκη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πόσο βραδικίνητη είναι η γραφειοκρατία του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Μιλάμε για μια οδηγία το 1991. Πολύ μεγάλο διάστημα αναμονής για απάντηση στη ανταπόκριση στις αλλαγές της αγοράς εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δύο πολιτικές ομάδες για το έργο τους και κάποιους που δεν συμμετέχουν στις ε, πολιτικές ομάδες, τους διερμηνείς που δύσκολη περίοδο ε, για αυτούς και τους σέβομαι ιδιαίτερα. Η δεύτερη ομάδα που ήθελα να ευχαριστήσω είναι αυτή ενώπιόν μου, οι φωτογράφοι, οι οποίοι εργάζονται υπό τεχνητό φωτισμό διαρκώς, είναι σημαντικοί, αλλά πολύ συχνά τους παραβλέπουμε. Ευχαριστώ λοιπόν τη φωτογραφική υπηρεσία για το έργο της. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μέγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορώ να υποστηρίξω αυτή την έκθεση. Οι εργατικοί οι βουλευτές μαζί με τους σοσιαλιστές και τους δημοκράτες ε, μαχήθηκαν για αυτούς τους νέους κανόνες που θα βελτιώσουν τις συνθήκες και θα δώσουν νέα δικαιώματα σε εκατομμύρια εργαζομένων που εργάζονται σε αβέβαιες συμβάσεις μηδενικών ορών. Έχω κουραστεί, έχω αιδιάσει να ακούω ανθρώπους να μου λένε ότι δουλεύουν σκληρά και δεν ξέρουν κάθε εβδομάδα αν τελικά θα έχουν αρκετά λεφτά για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αλλά έχει αρχίσει εντεπίθυση. Θα ε, σταματήσουν οι απολύσεις χωρίς αποζημίωση, να λαμβάνουν ειδοποίηση τελευταία στιγμή για νέες βάρδιες ε, χωρίς πληρωμή για ίση εργασία. Εμείς μαχόμαστε για να δημιουργήσουμε καλύτερες και δίκαιες συνθήκες εργασίας για τους πολλούς, όχι για τους λίγους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Μαριάς, παρακαλώ. Δίκαιε συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτουν την εφαρμογή τη ίδια τη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστή η Οδηγία 1999, η οποία διαμορφώνει συνθήκε προστασία όσων δουλεύουν με άτυπε μορφέ εργασία, όσων δουλεύουν με συμβάσει ορισμένου χρόνου και επιμένει η οδηγία αυτή του 1999 ότι θα πρέπει οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο βαθμό που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου και τέτοια κλασική περίπτωση είναι η περίπτωση της ομοιρίας των χιλιάδων ελλήνων δασκάλων οι οποίοι δουλεύουν με το σύστημα των αναπληρωτών και βρίσκονται όπως είπα σε ομοιρία και πρέπει επιτέλους το κράτος το ελληνικό να εφαρμόσει την οδηγία του 1999 και να διορίσει τους καθηγητές τους δασκάλους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως αναπληρωτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαμίκινς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλωσορίζω την οδηγία αυτή που ε, θέτει τα κατώτατα ε, δικαιώματα ε, που αφορούν όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι πολύ για τις λεπτομερές λίστες Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συνοριακή κινητικότητα μπορεί να δημιουργήσει εργαζομένους πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Απαράδεκτο για μένα, κατά τα άλλα. Ε, συμβάσεις εργασίας θα πρέπει να είναι αξιοπρεπής και να σταματήσει ε, ε, αυτή η επονίδιστη τακτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα έκανε ένα καλό βήμα που κατήργησε στο ιστορικό του Κοινοβουλίου τις άμυστες περιόδους άσκησης. Ε, θα πρέπει να προχωρήσει αυτό και στον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάουαρντ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά υποστήριζω αυτή την έκθεση. Είναι ένα σημαντικό πρωτοβήμα. Αναγνωρίζει το πρόβλημα της απασχόλησης μηδενικών μηδενικού ωραρίου. Είναι ένα πρώτο βήμα που διασφαλίζει ότι αυτές οι πρακτικές απασχόλησης θα τεθούν υπό έλεγχο ορθώς ζητάμε ίση μεταχείριση εργαζομένων ανεξαρτήτως της σύμβασης που έχουν υπογράψει. Ξέρουμε ότι η ευέλικτη οικονομία είναι μια πραγματικότητα και θα παραμείνει και συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα αυτών των ατόμων σε ε, πανευρωπαϊκό επίπεδο γιατί θα γίνει πανευρωπαϊκό το πρόβλημα αν δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν ζητάει κανείς πολλά όταν ζητά προβλέψιμες ώρες απασχόλησης και προβλέψιμα εισοδήματα από μια δουλειά δεν είναι παράλογο να μπορεί κανείς να υπολογίσει τα έξοδά του, να προβλέψει τα έξοδά του. Να σταματήσουν αυτές οι ανέλεκτες ώρες ε, ε, εργασίας και να απαιτείται από τον κόσμο να πληρώνει τη μαθητεία του. Αυτές, αυτά τα απαράδεκτα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Ευχαριστώ κύριο Σκαπού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι δημογραφικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων έχουν διαφοροποιήσει τον ενεργό πληθυσμό. Η ψηφιοποίηση έχει ευνοήσει νέες μορφές εργασίας υπαλληλικών σχέσεων με νέες σχέσεις εργασίας. Πιο ευέλικτες σήμερα μια σύμβαση εργασίας στις τέσσερις αντιστοιχείς, μόνο μια φορ... στις τέσσερις συμβάσεις αντιστοιχεί σε κλασική μορφή εργασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρώσεις τους θα έχουν το δικαίωμα να συμφωνήσουν με τον εργοδότη για τις περιόδους που είναι διαθέσιμοι και τις ειδοποιήσεις που μπορούν να δέχουν. Δεν θα μπορούν πλέον να απολυθούν, αν αρνηθούν να κάνουν μια δουλειά με ε, μία έγκαιρη προειδοποίηση και δεν θα μπορούν να δεχθούν ε, ωράρια, μηδενικά ωράρια. Δίνουμε σήμερα ε, το πράσινο φως για ένα νέο πυλόν εργασιακών δικαιωμάτων για την προστασία των πιο ευάλωτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη έκθεση, Λέναρς, ε, για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Το λόγο έχει η κυρία Σόεντροβα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εγώ ψήφισα υπέρ της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Παρά το γεγονός ότι δεν μου αρέσει να ε, ξεφυτρώνουν παντού νέε αρχέ, αλλά εγώ ψήφισα υπέρ. Διότι υπάρχει ανάγκη να παρακολουθούμε το κατά πόσο τηρούνται κάποιοι κανόνες ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά, η απόσπαση των εργαζομένων πρέπει να εφαρμόζεται σωστά το ίδιο και ολόκληρη η η νομοθεσία. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτή η αρχή εργασία, εργασίας, παρότι, την ονομάζουμε αρχή παρότι είναι περισσότερο ε, οργανισμός. Είναι σημαντικό λοιπόν τα καθηκοντά τη να μην επικαλύπτονται με τις αρμοδιότητες άλλων οργανισμών. Η υλοποίηση λοιπόν θα είναι σημαντική καθώς και ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θα ήθελα τα νέα κεντρικά τη ΕΛΕ να βρίσκονται σε ένα νέο κρατό μέλο. στη Σλοβακία θα ήθελα εγώ πιστεύω θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτή τη λύση. Ευχαριστώ κύριε Σπάλμερ. Είναι πάρα πολλοί αυτοί για τους οποίους ε, η οικονομία στι συντηρητικές κυβερνήσεις δεν λειτουργούν. Και το βλέπω αυτό στα Midlands καθημερινά. Ανασφάλεια εργασίες, συμφωνίε εργασίες ε, με μηδέν ε, ωράριο και μηδενικές ώρε να προβλέπονται και πολλά άλλα. Τίποτα χρήσιμο δεν θα έχουμε αν έχουμε κάτι να πούμε για τα θέματα αυτά. Είμαι υπερήφανο που σε αυτό το στο κοινοβούλιο ψήφισα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανασ... Ε, επισφαλούς εργασίας και την ε, απαγόρευση των ε, συμβολέων χωρίς προβλεπόμενο οργάριο. Σε λίγο οι ευρωβουλευτές, οι εργατικοί ευρωβουλευτές ε, θέλουν να συνεισφέρουν σημαντικά και επικοδομητικά στο χώρο αυτό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της αδικίας και της ανισότητας και θα εξασφαλίσουμε ε, ότι τα μέλη όλων των κοινοτήτων μας είτε ψήφισαν υπέρ ή κατά του Brexit ε, θα έχουν σοβαρή αντιπροσώπευση σε αυτό το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριος Δρογεύσκη. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μιλήσαμε για την κινητικότητα των εργαζομένων η οποία έχει διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της θητείας μας ακούγεται καλό, αλλά συνδέεται και με πολλά προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν κατά τη θητή αυτή, επαναλαμβάνω, και δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε επαρκώ αυτά τα προβλήματα. Αυτό ήθελα να τονίσω. Για την έκθεση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική μου ομάδα, το ΕΛΚΑ, για τη συνεργασία τους. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση, αλλά επικοδομητική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους μου και εδώ και στις Βρυξέλλες ε, και την Καμή για το άριστο έργο τους καθώς και το προσωπικό μου στο Βρότσφαφ στην Πολωνία τον Γιάννη Τσικόφσκι για παράδειγμα η Μόντρα θα ήθελα και τα δικά τους ονόματα να ακουστούν εδώ σε αυτή την αίθουσα γιατί αυτοί μου έδωσαν τη δυνατότητα να εργαστώ αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαριά. Okay. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να δρομολογεί την ίδρυση ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την εργασία καλό θα είναι κυρίως με την κομισιόν να κοιτάξει την εφαρμογή της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας και όσα κράτη παραβιάζουν την νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης για τα εργασιακά να τα παραπέμψει στο δικαστήριο. επανέρχομαι για πολλωστή φορά στην εφαρμογή της οδηγίας 1999 κάθετος 70 ε του Συμβουλίου και ζητώ την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας όπως είπα και σε προηγούμενες ομιλίες μου ζητώ την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας στην περίπτωση των αναπληρωτών δασκάλων. από τους 80.000 δασκάλους οι 20.000 είναι αναπληρωτές βρίσκονται σε ομοιρία τους εκμεταλλεύεται το ελληνικό δημόσιο και πρέπει επιτέλους να περάσει στο διορισμό τους δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται υπό πίεση προκειμένου να πετύχουν και την επόμενη χρονιά να επαναπροσληφθούν. πρέπει να υπάρξει οριστική ρύθμιση της περίπτωσης αυτής. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία είναι ένα μέτρο που περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό για να ολοκληρώσει τον κοινωνικό μα πλήλωνα. Τη χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να είναι εγγυημένη η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τα ίσα του δικαιώματα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, είναι απαράδεκτο να δρά ω απλώ μια θηρίδα ενημέρωση αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά ακόμα δεν μπορεί να βοηθάει τους πολίτες μας να λύνουν τα προβλήματα που έχουν με την εργασία τους. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία θα πρέπει να μπορεί να επιβάλλει τα μέτρα για να εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και να βεβαιώνεται ότι δεν προκύπτει νέα ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη νέα νομοθεσία. Και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στι χώρε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που ακόμα ε, έχουν οι συστήματα προστασίας ε, σε ό,τι αφορά την ανεργία και θα πρέπει να είναι στόχος της αρχής να εφαρμόζει τον κοινωνικό πυλώνα και να μην κλείνουν επιχειρήσεις και να μην χάνονται θέσεις εργασίας λόγω της εφαρμογής αυτών των νέων ε, διατάξεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαχραντήλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κοινωνική πολιτική είναι σημαντικός κλάδος ε, αρμοδιότητας των εθνικών κυβερνήσεων. Το ίδιο και τα, μας, τα κοινωνικά μας συστήματα. Γι' αυτό δεν ψήφισα υπέρ. Δεν διαφωνώ απλώς με την δημιουργία άλλου, ένα, ε, άλλου ενός ε, οργανισμού ευρωπαϊκού. Καταψήφισα διότι ανησυχώ ότι τέτοιοι οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα προσπαθήσουν να παρέμβουν σε ε, εργασιακούς νόμους και συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε κράτη-μέλη. Κάτι που πιστεύω υπερβαίνει κατά πολύ ε, το αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δουλειά της να παρεμβαίνει σε αυτά. Έχουμε 28 ε, και σύντομα 27 οικονομίες πολύ διαφορετικές, σχετικά εύπορες και σχετικά φτωχότερε χώρες. Δεν μπορούμε να τις βάλουμε όλες μαζί στο ίδιο πλαίσιο, στο ίδιο νομικό πλαίσιο. Θα ψήφισα κατά λοιπόν. Ευχαριστώ. Διακόπτε τη συνεδρίαση μέχρι τις 3. Γεια σας. Ευχαριστώ.